παρουσιάστηκε ωστόσο και θα ψηφιστεί την Τετάρτη. Είναι ένα ζήτημα πολύ σημαντικό η ανάπτυξη του Συμβουλίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Εθνών, συμπεριλαμβανομένου και του ρόλου τη ΕΕ, θα ψηφιστεί, επαναλαμβάνω. Προχωράμε λοιπόν αμέσω στην πέμπτη έκθεση, έκθεση για τα δημόσια οικονομικά τη ΟΝΕ κατά την περίοδο 2007 και 2008, ευθύνη τη βουλευτού κυρία Γκοτάρντι. Η κυρία Γκοτάλντι έχει το λόγο για τέσσερα λεπτά. Πρόεδρε, κυρία Επίτροπη, συνάδελφοι, πριν ένα χρόνο ακριβώ αναλάβαμε την, απο, την, λάβαμε την απόφαση να συνδέσουμε τις εκθέσεις για τα δημόσια των ετών 7 και 8 για δύο λόγους. Να πάμε πιο γρήγορα και να λάβουμε υπόψη τα ε, μηνύματα αλλαγών. Δεν ξέραμε βέβαια πόσο έντονες θα ήταν οι αλλαγές τότε, αλλά ξέραμε ότι, ήταν, ε, ότι αν, μπορούσαμε να αναλύσουμε, αν μπορούσαμε να αναλύσουμε τα δύο χρόνια θα είχαμε μια ε, πιο σφαιρική ανάλυση. Αυτό είναι αλήθεια. Η έκθεση βέβαια που ψηφίζουμε αύριο ενημερώνεται συνεχώ δεδομένων των στενών σχέσεων μεταξύ δημοσίων οικονομικών και οικονομική και χρηματοοικονομική κρίση. Αρκεί να σκεφτούμε το, τα κονδύλια που δόθηκαν για την διάσωση τραπεζών ή μεγάλων επιχειρήσεων, λαμβάνοντα υπόψη τα αιτήματα που, χωρίς να λάβουμε υπόψη τα αιτήματα που έθεσαν οι μικρομεσαίες επιχειρήσει και τις, τα, μέτρα που λαμβάνουμε για την προστασία των πολιτών από την ύφεση. Όλα αυτά ήταν θέματα που αφορούσαν και, τις, ε, και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα κράτη-μέλη, αλλά δεν θα έπρεπε να αποδυναμώσουν τι προοπτικέ και τι δεσμεύσει μα για το μέλλον. Η έκθεση περιλαμβάνει δύο επίπεδα το γενικό σταθερό επίπεδο που ισχύει σε κάθε επίπεδο και τις ανάγκες ε, αντιμετώπισης με κατεπίγοντα τρόπο της κρίσης. Είναι, ενισχύουμε την αρχή ότι ε, βιώσιμα δημόσια οικονομικά είναι απαραίτητα όχι μόνο για τα κράτη-μέλη αλλά και για την διατήρηση συνολικά της οικονομίας και του ευρωπαϊκού κοινωνικού μοντέλου. Σε ό,τι αφορά τις ε, ε, τα έσοδα, η μείωση της φορολογικής, του φορολογικής επιβάλλησης της εργασίας και των μικρομεσαίων ε, εισοδημάτων είναι το βασικότερο στοιχείο. Ταυτόχρονα, σε ό,τι αφορά τις δαπάνες, πρέπει να λάβουμε υπόψη τις ανάγκες του πληθυσμού, δίνοντας προσοχή στις πολιτικές φύλου και τις δημοκρατικές αλλαγές και όχι να κόψουμε δεν πρέπει να κόψουμε, να περικόψουμε αδιάκριτα, αλλά να, να, να, να διαμορφώσουμε τις δαπάνες, εξυγχρονίζοντας τα δημόσια οικονομικά. Μια χρήσιμη μεθοδολογία είναι αυτή του gender budgeting που το Κοινοβούλιο ε, προωθούσε εδώ και χρόνια, αλλά που ακόμα μακρόν, μακρά απέχει από την υλοποίησή της, παρά το ότι επιτρέπει την διαφάνεια, την συγκρισιμότητα, την γνώση από πλευρά των πολιτών και την αυξήσει την εμπιστοσύνη κατά συνέπεια και την αίσθηση ευθύνης. Η έλλειψη σταθερότητας πρέπει να αντιμετωπιστεί με σταθερούς τρόπους. Χρειάζεται παρέμβαση, είναι βασική παρέμβαση του δημόσιου τομέα, ωστόσο πρέπει να αποφύγουμε την επανάληψη παλαιών λαθών που είναι ακόμα πιο συγχώρητα τώρα και να εμποδίσουμε, και να εμποδίσουμε μια κρίση ε, που δεν θα είναι βιώσιμη. Όταν μιλάμε για την ανάγκη συντονισμού σε ευρωπαϊκό επίπεδο πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι αυτό είναι μια governance σε αντικυκλικό επίπεδο και με μόνο διάστατη προσέγγιση ε, αποφεύγοντας τη μάχη κατά της ε, καταπολεμώντας την, τους φορολογικούς παραδείσους και την φοροαποφυγή, λαμβάνοντας υπόψη τις επιπτώσεις των μέτρων στο, στην, στον ανταγωνισμό, τη λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, επιτρέποντας accountability, η αναθεώρηση των, του Συμφώνου σταθερότητα επιτρέπει ελεγχόμενη ευελιξία και πρέπει να την χρησιμοποιήσουμε με προσοχή και μακρόπνοα. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μακροοικονομικές πολιτικές κοινών επενδύσεων σε καθορισμένους εκ των προτέρων στρατηγικούς τομείς και να προσφέρουμε εργαλεία όπως αυτά των Eurobond, με δίνοντας μεγάλη προσοχή ταυτόχρονα στο υποεθνικό επίπεδο και στα περιφερειακά σχέδια σταθερότητας. Η έκθεση έτυχε ευρεία συνένεση στην Οικονομική Επιτροπή, δεδομένου το ότι οι περισσότερες πολιτικές ομάδες συγκλίνουν στην, ε, στην θέση που προ, και αυτό ελπίζω να είναι προάγγελος καλών αποτελεσμάτων στην αυριανή ψηφοφορία. Ευχαριστώ την Τονάτα. Κυρία Επίτροπε. President... Πρόεδρε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαιρετίζει <clears throat> την έκθεση Γκοτάρντι και η έκθεση αυτή ε, συμβαδίζει με δύο προηγούμενες ε, θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τον Ιούνιο του 2005 και του 2008 για τα δημόσια οικονομικά. Η έκθεση αυτή λέει, επιβεβαιώνει ότι το σύμφωνο σταθερότητας όπως αναπροσαρμόστηκε λειτουργεί καλά όπως θα έπρεπε. Πολλά κράτη-μέλη έκαναν ιδιαίτερες προσπάθειες για να ε, τηρήσουν τις υποχρεώσεις τους και μετά την μεταρρύθμιση ε, που έγινε τα πράγματα είναι καλύτερα οποιαδήποτε χαλαρότητα δεν δημιούργησε τα προβλήματα που φοβόντουσαν ορισμένοι από την άλλη μεριά οι προοπτικές για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ε, ζώνη του ευρώ είναι αρνητικές για το μέλλον η ανάπτυξη, ε, ο ρυθμός ανάπτυξης έχει μειωθεί σημαντικά. Μιλούμε για ύφεση ε, ενδεχομένως φέτος. Είναι αποθαρρυντικά τα πράγματα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν συμφωνεί με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι ε, μπορούμε να στηρίξουμε και να βοηθήσουμε τα πράγματα με ειδικά μέτρα δημοσιονομικής πολιτικής. Ε, από εκεί και πέρα βεβαίως είναι, ε, δεν μπορούμε να υπερβάλλουμε και γι' αυτό εμείς λέμε όπως λέτε και εσείς ότι η, τα δημόσια οικονομικά πρέπει να είναι βιώσιμα να μακροπρόθεσμα και τα τον, το φθινόπωρο του 2009 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα δημοσιεύσει μια έκθεση σχετικά με τη βιωσιμότητα των δημόσιων οικονομικών. Από εκεί και πέρα πιστεύουμε ότι οι δημόσιες δαπάνες θα πρέπει να αναπροσανατολιστούν ούτως ώστε να συμβαδεί αυθυγραμμιστούν με τη συνθήκη της Λισαβόνας. Κάτι τέτοιο είναι απαραίτητο και είναι με, αναφέρονται και στις κατευθυντήριες γραμμές του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Θεό. Πρέπει επίσης πρέπει να υπάρχει καλύτερη εποπτεία και παρακολούθηση της ποιότητας ε, των δημόσιων οικονομικών με βάση τις αρχές του performance budgeting. Αύριο θα ψηφιστεί και η έκθεση αυτή. Προχωρούμε τώρα στην έκθεση για τη μεταφορά στο εθνικό δικείο της, την εφαρμογή και την επιλογή της οδηγίας 2059 ΕΚ ε για τις αθέμετες εμπορικές πρακτικές των επιχειρήσεων προς τους κατανοητές στην εσωτερική αγορά και τις οδηγίες για την παραπλανητική και συγκριτική διαφήμιση